Καλησπέρα σας. Χθε και σήμερα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είχαμε φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά σήμερα το απόγευμα ξεκινάμε νωρίς. Είναι τιμή μας να έχουμε στο Προεδρείο την Επίτροπο Γιώχανσον για να μας ενημερώσει για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Εσωτερική Ασφάλεια. Τώρα υπεύθυνη είναι η επίτροπο Γιώχανσον, επίτροπο για τα εσωτερικά και για θέματα ασφάλεια. Ένα τομέα πολιτική που είναι σημαντικό για του Ευρωπαίου πολίτε, οπωσδήποτε, και βλέπουμε ότι οι επιλογές ε, υπόκεινται σε μια στρατηγική που έχει οριστεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου από τον Ιούνιο του 2015. Η στρατηγική κάλυπτε την περίοδο 2015 έως 2020 ως εκ τούτου, πράγματι χρειάζεται μια ενδελεχή συζήτηση για το θέμα αυτό. Η τρέχουσα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιστορική ασφάλεια περιλαμβάνει πολλά πολιτικά έγγραφα τα συμπεράσματα του 2014 του Συμβουλίου, την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, που προβλέπει την αντιμετώπιση τη τρομοκρατία και την πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση και στο διαδίκτυο, την ε, αναχέτηση του οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Έτσι, είχαμε και ένα ε, κοινό έγγραφο προεδρία τη Φιλανδική Προεδρία μαζί με τη Ρουμανική, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2019. Εδώ ε, θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Γιώχανσον για το θέμα, τις πρόσφατες εξελίξεις ε, στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και το μέλλον. Το μέλλον που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Ο προβλεπόμενος χρόνος για αυτή την ανταλλαγή απόψεων είναι μία ώρα να το έχετε παρακαλώ υπόψη, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε σε λογικά πλαίσια. Έχετε το λόγο, Επίτροπε Γιώχανσον, για τα επόμενα 10 λεπτά. Και μετά θα έχουμε ένα πρώτο γύρο συντονιστών. Για του συναδέλφου που θέλουν να πάρουν μέρο στη συζήτηση, παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σα, τι καρτέλε σα. Τέλο πάντων, φροντίστε να σημειωθείτε στον κατάλογο. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και θα μιλήσω για την εσωτερική ασφάλεια. Για μένα η εσωτερική ασφάλεια και η ελευθερία είναι αλληλένδυτες. Το θέμα είναι η συνοχή στην κοινωνία και πώς οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται ελεύθεροι να δράσουν ε, όπως και οι άντρες. Πώς τα παιδιά ε, θα προστατεύονται, γιατί έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε βία η ενέργεια ή κακοποίηση. Υπάρχουν πολλές λοιπόν σοβαρές πτυχές της εσωτερικής ασφάλειας. Όπως όλοι γνωρίζετε, ε, εξαρτώμαθα ημένα από τους ΔΕ για την ασφάλεια των άλλων. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε. Γνωρίζουμε ότι παρόλο που είχαμε θετικές εξελίξεις, η εμπιστοσύνη ενισχύεται μεταξύ των κρατών μελών, αλλά έχουμε ακόμα πολλά μπροστά μας να κάνουμε. Έχουμε βελτιώσει τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε απειλές κατά της εσωτερικής ασφάλειας, όμως το έγκλημα κινείται και στο διαδίκτυο. Αναπτύσσονται νέα τεχνολογικά μέσα και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, για να το πω έτσι. Πριν περάσω στις νέες μας προτάσεις, πρώτα Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε μια απόφαση που ήδη έχουμε λάβει, ιδίως την υλοποίηση των νέων συστημάτων επικοινωνίας για την διαλογικότητα. Ρωτήσαμε τα κράτη-μέλη πώς ε, θα ε, περάσουν στη δηλοποίηση και αν είναι προετοιμασμένα και έχουν ακόμα πολλά να κάνουν. 16 κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα εθνικό πρόγραμμα υλοποίησης. 11 κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα κάνει αξιολογήσεις της εθνικής του νομοθεσία ή αυτής που λείπει και 12 δεν έχουν καν εκτίμηση των πόρων που θα απαιτηθούν. 17 ε, κρατη δεν έχουν λεπτομερές πρόγραμμα. Αυτό ήταν ένα από τα μηνύματά μου την περασμένη εβδομάδα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών. Ότι ο κάθε υπουργό θα πρέπει να φέρει ε, στην πρώτη θέση ε, το θέμα αυτό. Επαφιόμαστε στο καθένα κράτος μέλος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα αυτά μέχρι να κάνει ο τελευταίος όσα πρέπει για να υλοποιηθούν. Πρέπει να βιαστούν. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό για μένα και θα το παρακολουθώ. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι η πρόταση που εκκρεμεί για το τρομικό, τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και το e-evidence, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Με το νέο κοινοβούλιο τώρα έχουμε και νέου εισηγητή και σκιώδει εισηγητέ. Πρέπει λοιπόν αυτό να το προωθήσουμε και σε πολιτικό επίπεδο. Είμαι έτοιμη να συνεργαστούμε για να βρούμε μια συμβαστική λύση σε συνεργασία με το Συμβούλιο για τη διασυνεργειακή διάσταση ε, του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Γιατί και τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Επίση, ε, το νομοθέτημα για τι ηλεκτρονικέ ε, αποδείξει είναι σημαντικό γιατί 85% των ποινικών υποθέσεων και ερευνών περιλαμβάνουν και συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Να πω τώρα κάτι για την νέα πρόταση, τι νέε πρωτοβουλίε που προγραμματίζω. Αλλά πριν περάσω στι λεπτομέρειε, να πω ε, ότι σε ό,τι αφορά την προετοιμασία νέας νομοθεσίας είμαι ε, έτοιμη να ε, διασφαλίσω ότι θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, πραγματικά και απτά στοιχεία για μετά από διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους και μελέτες αντικτύπου όσο το δυνατόν περισσότερο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Πρέπει να προετοιμάσουμε τις νέες προτάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι τρει ε, τομεί προτεραιότητα θα είναι ε, η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, το, το, οργανωμένο, το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Με συγχωρείτε. Και η καταπολέμηση του ε, εγκλήματο στην ψηφιακή εποχή. Σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση, έχουμε ήδη κάνει πολλά, όπω είπα, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Έχουμε δει ότι περίπου όλες οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν διαπραχθεί από, όπως λέγονται, τρομοκράτες που έχουν μεγαλώσει εδώ, στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ε, χαρακτηριστικό είναι ότι χρησιμοποιούνται μέσα χαμηλού κόστους και χωρίς ιδιαίτερη τεχνολογική ε, ε, εξέλιξη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να ανοιχετήσουμε και, σε, και αυτές τις ενέργειες. Επίσης υπάρχουν νέες απειλές με ε, χημικές ουσίες, με μη επενδρομένα αεροσκάφη. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλα τα ευπαθή σημεία του διαδικτύου που μπορεί να εκμεταλλευτούν οι τρομοκράτες για τους, σκοπού, για τους σκοπούς τους. Η τρομοκρατία των τσιχαντιστών παραμένει μια σοβαρή απειλή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως υπάρχουν και άλλες απειλές από τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές Κατά τα στοιχεία της Europol έχουμε 129 αποτυχημένες επιθέσεις από το 2018, οι επιθέσεις που αναχαιτίστηκαν. 56 άτομα συνελήφθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια αδικήματα την ίδια χρονιά. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την αστυνομική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και πρέπει να έχουμε αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα αλλά και να εντοπίζουμε τους ξένους μαχητές που μπορεί να θέλουν να επιστρέψουν. Πρέπει να κάνουμε και περισσότερα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση κατά της ριζοσπαστικοποίησης συμπεριλαμβάνει ε, ειδικού και ανθρώπου που εργάζονται στην πράξη με τα θέματα αυτά, καθώ και νομικού, αλλά θα περάσουμε μετά σε περισσότερε λεπτομέρειε για το δίκτυο αυτό. Θα συνεχιστεί και ο διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, διότι υπάρχει το Φόρουμ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ιντερνετ, που έχει αποδειχθεί μια πολύ ε, πολύτιμη οδό για να ε, συνεχίσουμε την ευαισθητοποίηση για το επικίνδυνο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε νέε προτάσει ό,τι αφορά τι κρίσιμε υποδομέ. Σήμερα η νομοθεσία περιορίζεται στην ενέργεια και τις μεταφορές μόνον. Είμαστε ε, στη φάση που προετοιμάζουμε προτάσεις ε, για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ε, υγειονομικούς καθώς και την διαχείριση των υδάτων, την Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, πρέπει να επιταχύνουμε την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο. Βάσει των στοιχείων τη Europol, 5.000 οργανωμένε ομάδε αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται υπό ε, έρευνα στην Ευρώπη. Έχουμε αύξηση περίπου 50% σε σχέση με το 2013. Πρέπει να βελτιώσουμε την αστυνομική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Και αυτό φυσικά είναι ιδιαίτερα σκόπιμο για την καταπολέμηση και τη τρομοκρατία. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε τη συνεργασία των διοκτικών αρχών και το πλαίσιο τη, γιατί για την αστυνομία χρειαζόμαστε και ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για να συγκεντρώσουμε απερχιωμένα και διασκορπισμένα σε διάφορα νομοθετήματα νομικά κείμενα, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν ε, αποτελεσματικότερα. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε την εντολή της Europol. Θα πρέπει ο οργανισμός να είναι σε θέση να ανταλλάσσει στοιχεία απευθείας με ιδιωτικές εταιρείες όπως τράπεζες για ποινικά δικήματα ή ε, οργανώσεις για τις περιπτώσεις τρομοκρατίας παιδικής πορνογραφίας. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που οι διεκτικές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες, κοιτάζοντας ποια είναι η πηγή ε, της έρευνας, με τις αποφάσεις προύμ, όπως λέγονται. Ε, με αυτές θα μπορούν τα κράτη-μέλη να ψάχνουν απευθεία ε, την καταγραφή των οχημάτων, τα δακτυλικά αποτυπώματα, το γενετικό υλικό, όπως έχουν καταγραφεί στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Όμως αυτά δεν είναι επικαιροποιημένα. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις δυνατότητες ανταλλαγής στοιχείων και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν νέε κατηγορίε στοιχείων και να βρούμε νέου τρόπου διαλογικότητα ε, και διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων. Είναι τεράστιοι οι πόροι που διαθέτουν οι ομάδε οργανωμένου εγκλήματο. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τι δυνατότητε παγώματο και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα μόνο 1% αυτών των εσόδων που παράγει το οργανωμένο έγκλημα μπορούν να κατασχεθούν. Είναι ένα τομέα όπου χρειάζεται να έχουμε νέε προτάσει για να πάψει η ροή ρευστού θα πρέπει να πάψει και η εμπορία ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά δεν είναι μόνο απειλή κατά των ε, ατόμων και των οικογενειών, αλλά πραγματικά είναι και πηγή εσόδων για το οργανωμένο έγκλημα. Βλέπουμε περισσότερα ναρκωτικά φτηνότερα και δυνατότερα, ε, τα οποία ε, κυκλοφορούν και παράγονται και στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να υποβάλουμε μια, ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τα ναρκωτικά και την καταπολέμησή του. Θα παρουσιάσω και ένα πρόγραμμα δράση για την εμπορία των πυροβόλων όπλων. Τα παράνομα όπλα δίνουν δυνατότητε τη ομάδα οργανωμένου εγκλήματο και στου τρομοκράτε που μπορούν να διαπράξουν εγκλήματα. Βάσει μια μελέτη το 2018, 35 εκατομμύρια παράνομα πυροβόλα όπλα βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων επίση. Θέλω να ε, να μην υπάρξει ατιμορρησία για τον οποιονδήποτε εμπλέκεται στην αλυσίδα της εμπορίας και να πάψει αυτή η αποποινικοποίηση όσων έχουν κάποια εμπλοκή. Θα πρέπει να, μην, υπάρξει μεγαλ... να μην υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες από την πλευρά των εγκληματιών, αλλά να ενισχύσουμε τους, ε, τις διοκτικές αρχές. Η τεχνητή ευφυΐα, τα ψηφιακά μέσα δίνουν νέες δυνατότητες. Θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και εμείς από την πλευρά μας. Σήμερα οι διοκτικές αρχές χάνουν τη μάχη για την προστασία των παιδιών που ε, πέφτουν θύματα κακοποίηση στο διαδίκτυο. Αυτό το σοβαρό έγκλημα έχει διωγγωθεί και ε, γνωρίζει, για να το πω έτσι, άνθηση. Οι αστυνομικοί μα θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα αποτελεσματικότερα και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα οι παραβάτες ε, με σεξουαλικά εγκλήματα κατά των παιδιών, εις βάρος παιδιών, ε, εκμεταλλεύονται το ανώνυμο που τους προσφέρει το διαδίκτυο, καθώς και τις δυνατότητες κωδικοποίησης δεδομένων. Μπορούν έτσι να αποθηκεύουν και να μοιράζονται περιεχόμενο, χωρίς να μπορεί εύκολα να τους εντοπίσει κανείς. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα των υποεξέλιξη ερευνών. Το κέντρο για το κυβερνοέγκλημα της Europol ε, ε, υπολογίζει ότι έχουμε τουλάχιστον 200.000 ενεργούς χρήστες σε πλατφόρμες με ε, υλικό που χρησιμοποιούν την κωδικοποιημένη του ταυτότητα για να μπορούν ε, να κρύβουν ε, υλικό που έχει σχέση με παιδική πορνογραφία. Είναι σημαντική αυτή λοιπόν η δράση ε, μεταξύ των νέων μας πρωτοβουλειών. Εν είδη συμπεράσματος πολλά έχουμε επιτύχει ήδη, αλλά νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και τα κράτη-μέλη και ιδίω εσείς, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, Περιμένετε να κάνουμε ακόμη περισσότερα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, να προστατεύσουμε τις γυναίκες, τα παιδιά και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών της κοινωνίας γενικότερα και μεταξύ των κρατών μελών. Είμαι πεπισμένη ότι αν συσπηρωθούμε και εργαστούμε σκληρά ε, σε συνεργασία όλων των κρατών μελών μεταξύ τους και των ε, αρχών που είναι υπεύθυνε για την ασφάλεια, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Περιμένω με ανυπομονησία τις ερωτήσεις σας και τις συνεισφορές σας για τις νέες προτάσεις που σκέφτομαι να υποβάλω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την επισκόπηση των ε, θεμάτων που μας ενδιαφέρουν. Να ξεκινήσουμε από τους συντονιστές ε, και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο να σηκώσουν το χέρι τους ε, για να τους καταγράψουμε στον κατάλογο των ομιλητών. Πιατσόλα, Μετσόλα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που επανήλθατε στην Επιτροπή μας ε, για να έχουμε επικοδομητικό διάλογο πάνω στα θέματα ενδιαφέροντός μας. Όταν μιλάμε για την ζώνη Σέγγεν και την έλλειψη εσωτερικών συνόρων είναι κάτι ε, το οποίο ε, το επενούμε και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αλλά θα θάβαμε το κεφάλι μας στην άμμο εάν δεν καταλαβαίναμε ότι υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες ως προς την ασφάλεια διότι η δυνατότητα αυτή ε, ε, αποτελεί ε, αντικείμενο εκμετάλλευσης και από εγκληματίες για σκοπούς τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε ότι τα ασφαλή εξωτερικά σύνορα αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του Σέγγεν. Πώς μπορούμε ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αυξήσουμε τα μέτρα στα σύνορά μας για να διασφαλίσουμε την εσωτερική μας ασφάλεια. Επίσης θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας με τρόπο σωστό και αναλογικό. Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα κράτη-μέλη, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς βλέπετε τις δυνατότητες βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και επίσης αναφερθήκατε στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας αυτή ήταν μια πολύ ε, δύσκολη διαδικασία. Σας καλώ να φροντίσετε όλα τα κράτη-μέλη αλλά ε, και ενδιαφερόμενοι φορείς ε, να ε, συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαβούλευση όπως είναι για παράδειγμα οι συλλέκτες και οι αθλητές διότι το θέμα των πυροβολών όπλων έχει να κάνει όχι μόνο έχει να κάνει με δραστηριότητες στα κράτη-μέλη που δεν είναι πάντα εγκληματικές. Ε, πρόεδρος, ε, συνάδελφοι, το πρωί είχαμε καθυστέρηση ε, επειδή είχαν συσσωρευτεί διάφορα θέματα και διάφοροι συνάδελφοι ήθελαν να πάρουν το λόγο. το ίδιο ισχύει τώρα και το απόγευμα. Έχουμε πάνω από 20 ανθρώπους στον κατάλογο των ομιλητών. προτείνω να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε, ε, να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα, ε, οι συντονιστέ δηλαδή να έχουν από δύο λεπτά, οι υπόλοιποι ευρωβουλευτέ από ένα λεπτό για να θέσουν τι ερωτήσει του. Ε, συμφωνείτε, σα παρακαλώ να μα στηρίξετε, διότι αλλιώ πάλι θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Η κυρία Σίπελ, σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή και για τον διάλογο αυτόν. Σήμερα το πρωί είχαμε ανταλλαγή απόψεων ε, στην αύξηση, ε, είχαμε συζήτηση πάνω στην αύξηση της εισαγωγής ναρκωτικών σε μεγάλα κοντέινερ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ λοιπόν ότι ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων είναι υψηλής της σημασίας αλλά επιλέγουμε να ενισχύσουμε τον Frontex, να ε, ε, ενισχύσουμε την ε, συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Κατά την εφαρμογή και επιβολή του νόμου όμως έχουμε καθυστέρηση, διότι τα κράτη-μέλη δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα στην πράξη. Ακούσαμε τα στοιχεία σχετικά με τη διαλειτουργικότητα. Ακούσαμε ποιες ή πόσες χώρες αρχίζουν να εφαρμόζουν ε, τα σχετικά μέτρα και πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση από πλευρά των κρατών μελών. Αναρωτιέμαι λοιπόν, χρειαζόμαστε πράγματι νέα μέτρα ή πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην εφαρμογή των μέτρων που ήδη έχουμε θεσπίσει ή μή, οι αποφάσει μας έχουν καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την εφαρμογή τους. Ακούσαμε επίσης ότι το, ε, στο οργανωμένο έγκλημα ε, υπάρχει πολύ γρήγορη προσαρμογή σε νέε ε, ευκαιρίες ε, και ε, αλλαγής κατεύθυνσης. Πέρα λοιπόν από όλα τα μέτρα, μπορεί ο τομέας επιβολής του νόμου να φροντίσει να έχει εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς αυτούς. Ε, θα πρέπει οι εθνικέ μα αρχέ να ασχοληθούν με αυτό, ώστε να έχουν εξειδίκευση του προσωπικού του και να έχουν εμπειρογνώμονε στου διάφορε τομεί, ομάδε εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση των διαφόρων ειδών εγκλήματος. Ε, πριν λίγο καιρό αστείευτηκα, αλλά ίσω τελικά να είναι καλή ιδέα, να έχουμε κάτι σαν ε, πρόγραμμα Εράσμου στον τομέα επιβολή του νόμου, ώστε να μπορεί να γίνεται ανταλλαγή απόψεων εμπειριών, να μαθαίνει ο ένα από τον άλλον για να αντιμετωπίζονται καλά οι προκλήσει όλων των κρατών μελών. Πιστεύω ότι όλοι συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί με περισσότερες μορφές συνεργασίας, περισσότερες κοινέ ερευνητικέ ομάδες, ώστε να μπορεί να βελτιωθεί και η κατανόηση του προβλήματος πέρα από την λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Επίση, μιλήσατε για την άνοδο του εξτρεμισμού και εγώ που είμαι Γερμανίδα ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από την τρομοκρατία όσον αφορά την απειλή προς την τρομοκρατία διότι όσον αφορά την εξωτερική τρομοκρατία όλοι λένε ναι αυτό είναι απαράδεκτο πρέπει να το καταπολεμήσουμε αλλά διάφορες μορφές εξτρεμισμού ε, απειλούν τη δημοκρατία μας διότι όλο και περισσότεροι απειλούνται, οι οικογένειε τους απειλούνται και πολύ συχνά δεν έχουν ε, το θάρρος να ε, προσφύγουν στις ε, αρχές και ε, βλέπουμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αδράνεια και αυτό απειλεί την ευημερία των ανθρώπων. Τέλος, κυβερνοασφάλεια και όλα τα εγκλήματα στο διαδίκτυο. Πιστεύω ότι είναι θλιβερό ότι πάντα αναφέρουμε την ε, ε, κακοποίηση ανηλίκων σε αυτό το πλαίσιο. Πράγματι είναι πρόβλημα. Ε, η κρυπτογράφηση όμως είναι υψίστης σημασίας και θα ήθελα να δω τι ακριβώς κάνουμε, διότι λέμε ότι αυξάνεται η κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο. Ε, ειλικρινά, οι φωτογραφίες και τα ζωντανά βίντεο που δείχνουν ε, πραγματοποιούνται και στην πραγματική ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται στην πραγματική ζωή και όχι μόνο ε, να κυνηγάμε τις φωτογραφίες. Ναι, πράγματι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Σήμερα το πρωί ε, χρειάστηκε να ζητήσουμε παράταση από τους ε, διερμηνείς. Ε, μου φαίνεται ότι και σήμερα, ότι και τώρα το απόγευμα θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό. Ε, ή να συνεχίσουμε τη συζήτηση στα αγγλικά. Όπως και να έχει, θα είναι χρήσιμο εάν οι συντονιστές περιοριστούν στα δύο λεπτά και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές σε ένα λεπτό, διότι 25 ομιλητέ έχουμε. Ήδη έχουμε ε, καθυστερήσει ως προς το χρονοδιάγραμμά μας. Σας παρακαλώ λοιπόν βοηθήστε κι εσείς. Η κυρία Ινετφέλτ. Θα είμαι σύντομη. καλώ ήρθατε κυρία Επίτροπε στην Επιτροπή μας. Είπατε ότι από εδώ και στο εξή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει πολιτικές που να βασίζονται σε στοιχεία. Το καλωσορίζω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι σε σχέση με το παρελθόν και άρα θα υπάρχουν προτάσεις οι οποίες δεν θα καταπίπτουν εκ των υστέρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καλό θα ήταν αυτό. Ή επίσης θα λάβετε υπόψη σας τις σχετικές συστάσεις της ε, ε, Αρχής Θεμελιωδών Ελευθεριών και του ε, Επόπτη Δεδομένων. Επίσης, φαντάζομαι ότι θα λάβετε υπόψη σας ε, πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή, γιατί γρήγορα υιοθετούμε νέα νομοθετήματα, αλλά είναι τραγική η εφαρμογή τους. Και ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, η Λίμπε επισήμως να μπορέσει να ζητήσει, όπως συμβαίνει στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, να έχουμε, να δημιουργήσουμε ένα βαθμολόγιο της ε, εφαρμογής της ε, νομοθεσίας για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για να κοιτάμε πώ θα πηγαίνει η Επιτροπή. Γιατί, για παράδειγμα, από το 2009 ήταν υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη να προμηθευτούν ε, το, τους, το μηχανήματα που χρειάζονται για να λαμβάνουν κτηλικά αποτεπώματα για να τα βάζουν στα διαβατήρια. Και 11 χρόνια μετά, μόνο 9 κράτη-μέλη έχουν προμηθευτεί το σχετικό εξοπλισμό. Και τι κάνει η Επιτροπή, Επίση, πολύ σπάνια και λίγα πράγματα ακούω από την Επιτροπή για ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Σε αυτή λοιπόν την οδηγία θα μπορέσει να με ενημερώσει για την Ελλάδα, για την Ισπανία, για την ε, Σλοβενία, οι ε, οποίες, κατά των οποίων ε, έχετε ξεκινήσει διαδικασία επί για το γεγονό ότι δεν έχουν Ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο την σχετική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιούν ακόμα την οδηγία πριν το 2008, δηλαδή πριν το iPhone. Επίσης, συχνά αναφερόμαστε στην τρομοκρατία. Όμω ας μιλούμε και για, ξεκάθαρα για την ακροδεξιά τρομοκρατία ή επίσης για τη βία κατά των γυναικών. Γιατί εάν έχουμε χιλιάδες ε, ε, ε, γυναίκε να πεθαίνουν από τη βία κατά των γυναικών στην Ευρώπη κάθε χρόνο, αυτό δεν είναι πια ιδιωτικό ζήτημα. Επίση, 10 δευτερόλεπτα για να κλείσω. Καλωσορίζω την πρότασή σας να επικαιροποιηθεί η εντολή, αλλά όχι μόνο για να έχουμε την δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επίσης για τον έλεγχο και των διοκτικών αρχών, γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη διαπιστώνουμε, την εντολή τη Europol λοιπόν, να ε, διαπιστώνουμε οι ίδιε οι κρατικέ αστυνομικέ αρχέ να είναι διεφθαρμένε. Και αν ε, δεν γίνει αλλαγή τη εντολή τη Europol για να μπορεί να το διαρευνά και αυτό, δεν θα προχωρήσουμε. Και επίση θα πρέπει και η Europol να αποκτήσει του κατάλληλου πόρου που χρειάζεται για να τα καταφέρνει όλα αυτά. Για τους πράσινους, η κυρία Στέκ, εγώ θα κρατήσω τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την γενική επισκόπηση των προτεραιοτήτων σας. Καλωσορίζουμε την προσέγγιση που λέτε ότι θα έχετε, δηλαδή ότι θα γίνεται μια αξιολόγηση αντικτύπου εκ των προτέρων πριν προτείνεται νέα νομοθεσία και ότι αυτή θα βασίζεται σε στοιχεία. Ελπίζουμε ότι αυτέ οι αξιολογήσει αντικτύπου θα εξετάζουν κατά πόσο χρειάζεται στην πραγματικότητα αυτή η νομοθεσία ή μήπω εάν υπάρχουν ήδη εργαλεία που θα κάλυπταν το θέμα και επίσης ότι θα εξετάζεται εάν θα είναι συμβατή αυτή η νομοθεσία με ε, υφιστάμενα πρότυπα, όπως για παράδειγμα την προστασία προσωπικών δεδομένων, γιατί μιλούμε για παράδειγμα εδώ για ανταλλαγή δεδομένων, ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι ε, συμβατό, θα γίνεται με τρόπο συμβατό με την νομοθεσία και την ομολογία. Έχουμε νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, η Σύμβαση τη ε, Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν την έχουν κυρώσει ακόμα και αναρωτιέμαι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διορθώσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το κενό. Συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη αμοιβέ εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι σιγά σιγά μειώνεται, εάν, εάν μάλλον ε, κοιτάξουμε τι προβλήματα με το κράτος δικαίου υπάρχουν σε κάποια κράτη και τι κάνουμε γι' αυτό. Επίση, λέγεται ότι μπορεί, μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, εναρμόνιση τη νομοθεσία για τα διαδικαστικά εχέγγυα τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό. Επίση, για το νέο θεματολόγιο για τα ναρκωτικά που μα λέτε. Ελπίζω να λάβετε υπόψη σα και το γεγονό ότι υπάρχουν διαφορετικέ πολιτικέ, διαφορετικέ προσεγγίσει στην πολιτική για τα ναρκωτικά μεταξύ κρατών μελών. Και ίσω σε ορισμένε περιπτώσει η νομιμοποίηση να είναι πιο αποτελεσματική. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κέρδο που αντιπροσωπεύουν τα ναρκωτικά για τι εγκληματικέ ομάδε και να είναι μια τελικά πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Επίση, λέτε ότι θέλετε να ενισχύσετε την συνεργασία αντί για νέα νομοθεσία. Για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες. Η Europol, η Eurojust δυστυχώς συνεχίζουν να βασίζονται στα διαρθρωτικά ταμεία. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τι πόρους τους δίνουμε και σε ανθρώπινους πόρους και σε οικονομικού πόρου και τι μπορούμε να συνεισφέρουμε εθνικά και ευρωπαϊκά για να μπορούν με τρόπο προβλέψιμο να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους έχουμε αναθέσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κ. Σταντίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Οι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική αναφέρθηκαν από την Επίτροπο Τρομοκρατία κατά πολέμηση της, ε, του οργανωμένου εγκλήματο στο διαδίκτυο, και σοβαρέ οργανωμένε εγκληματικέ ομάδε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στη διασυνοριακή διάσταση για την, την εμπορία ανθρώπων, την πορνεία, την τρομοκρατία και την διακίνηση ναρκωτικών. Από το 2011 έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, αλλά απέχουμε πολύ από την πραγματικά δραστική αναχέτηση που να δώσει μια τελική λύση στο πρόβλημα. Για να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά, χρειάζεται καλύτερη δικαστική συνεργασία και των αστυνομικών αρχών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορέ μεταξύ των περιοχών τη Ευρώπη και σε εθνικό επίπεδο και να υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 100 μελών. Οι καθημερινέ ειδήσει μα δείχνουν ότι παρά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και του στρατηγικού μα στόχου, ακόμα είμαστε πολύ ευπαθεί. Οι επιθέσει που έχουμε δεχτεί το αποδεικνύουν ο αυξανόμενο ρυθμός ε, των τεχνολογικών εξελίξεων δυσκολεύει την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών στο διαδίκτυο με ψηφιακά μέσα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. Όπω ξέρετε, στι συζητήσει που γίνονται στο Συμβούλιο για τη μελλοντική εξέλιξη τη ιστορική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οργανωμένο έγκλημα προκύπτει λόγω τη ζήτηση και τη προσφορά ευκαιριών στι ε, εταιρείε που δρούν εγκληματικά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια της πολιτικής μας όπως αυτή των ανοιχτών λιμένων. Ε, γιατί η ασφάλεια φτάνει στα όρια της, ιδίως στην Αφρική. Ριζοσπαστικοποίηση βίαιη πολλές φορές υπάρχει στην Ευρώπη και είναι μια απειλή από, κατά της εσωτερικής μας ασφάλειας. Για αυτά τα θέματα, Επίτροπε, ήθελα να μου πείτε αν πραγματικά υπάρχει κάποιο απτό σοβαρό πρόγραμμα πέραν των γνωστών προγραμματικών δηλώσεων, τις οποίες τις ακούσαμε και είναι πολύ ευχάριστε να τι ακούμε μεν, αλλά κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε. Συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ, ο κύριο Προκατσίνη. Δεν είναι εδώ. Η κυρία Κάνκο. Ναι, όχι. Βλέπω το όνομά σας. Εσείς, για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ή εσείς κυρία Κάνκο. Κυρία Κάνκο, έχετε το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Um, Σας ευχαριστώ που τονίσατε τα σημαντικά αυτά θέματα ιδιαίτερα. Ε, μ' αρέσει το ότι θα υπάρχει δυνατότητα αυξημένης ανταλλαγής ε, δεδομένων ε, και με την Europol. Εγώ έχω ερώτηση σχετικά με την έντολη του Frontex. Νομίζω ότι μετά από όλες τις ανακοινώσεις και τη δημοσιότητα στο θέμα αυτό μετά τις 4 Δεκεμβρίου νομίζω ότι θα πρέπει ο οργανισμός αυτός να παρουσιάσει αποτελέσματα, διότι όταν ε, μας ε, ρωτούν ε, οι πολίτες τι έχουμε να τους πούμε, δεν είναι τίποτα σαφές αυτή τη στιγμή. Η νέα εντολή θα διασφαλίσει καλύτερες επιστροφές, καλύτερο έλεγχο των συνόρων. Μία πτυχή της εντολής είναι η επανένταξη των επιστρέφοντων σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πολιτική μετανάστευση είναι σημαντικό όμως και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, από την ε, εκμετάλλευση και η προστασία αποτελεί σημαντική πτυχή των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών για να αυξηθεί και η ε, εμπιστοσύνη του κοινού. Ποιε είναι οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού επιστροφής σε τρίτες χώρες Ιδιαίτερα πολλές γυναίκες και κορίτσια βρίσκονται στην ε, θέση αυτή και ε, θα επωφεληθούν από μια καλή πολιτική επιστροφών. Ευχαριστώ από την ΚΟΕ η κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις σε τρεις τομείς για το σύστημα πληροφόρησης Schengen, ε, ιδιαίτερα ε, δεδομένης της ε, αντιγραφής των βάσεων δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, παραβιάζοντας τους κανόνες που έχουν επιβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εφόσον δεν ήταν μέλος του Σέγγεν. Ρωτώ λοιπόν γιατί δεν υπήρξε διαδικασία επιπαραβάση για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και ο μηχανισμός παρακολούθησης που εντόπισε αυτές τις παραβιάσεις γιατί ε, ανεστάλλει η λειτουργία του και ε, αφότου διαπιστώθηκαν αυτές οι παραβιάσεις, ε, τι έγινε με τις βάσεις δεδομένων που είχαν αντιγραφεί παράνομα και τι έγινε με τους ανθρώπους των οποίων τα δεδομένα έτσι δόθηκαν χωρίς άδεια. Και ερωτώ επίσης Τώρα που θα είναι ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, τι θα γίνει με τα ευαίσθητα αυτά δεδομένα, ε, συχνά αφορούν και DNA. Υπήρχαν και άλλα προβλήματα από άλλες χώρες όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων για τις θεωρήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο ήταν οι δυνατότητες υποκλοπής δικτύων 5G στο πρότυπο 5G υπάρχει μηχανισμός κυβερνοασφάλειας, ο οποίος όμως ε, φαίνεται ότι ε, παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά τις υποκλοπές. Ε, εσείς τι εννοείτε εσείς ε, τι πιστεύετε, πώς θα αλλάξετε ε, τα πρότυπα του 5G ε, όσον αφορά την ασφάλεια και στην πράξη τι ζητάτε από τους παρόχους δικτύου να κάνουν. Και επίσης όταν μιλάτε για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού δεν συμφωνείτε ότι ο καλύτερος τρόπος να γίνει ασφαλής η Ευρώπη είναι να σταματήσουμε να παρεμβαίνουμε σε κυρίαρχες περιοχές στη Μέση Ανατολή και αλλού ε, διότι αυτές είναι οι προϋποθέσεις ε, που οδηγούν ε, στον εξτρεμισμό και στην βία. Ευχαριστώ. Κυρία Ιωχάνσον, προτείνω να δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές, ένα λεπτό στον καθένα. Ένα λεπτό ο καθένας για να μην ξεπεράσουμε το χρόνο μας. Ένα λεπτό, κύριε Σαρθαλέγκος. Ευχαριστώ πολύ. Την ε, προηγούμενη ε, εβδομάδα ο, ο, η αντιπρόεδρος της ε, Βενεζουέλας εισήλθε σε ευρωπαϊκό έδαφος κατά παράβαση των κυρώσεων. Προσγειώθηκε στην Μαδρίτη και συναντήθηκε με εξέχον στέλεχος της Ισπανικής κυβέρνησης έκτοτε. Έχει αναφερθεί το θέμα αυτό αρκετέ φορέ. Ο ε, ε, υψηλό εκπρόσωπο όμω είπε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν ε, τι κυρώσει. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω αν γνωρίζετε εσεί αυτήν την παράνομη είσοδο παραβιάζοντας ε, τις ευρωπαϊκές κυρώσεις από τον Αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας ε, και ε, είσαστε διατεθειμένοι να ζητήσετε πληροφορίες από την Ισπανική κυβέρνηση για να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό, το οποίο επηρεάζει το σύνολο του καθεστώτος κυρώσεων που αφορά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Έλισετ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, εισήγηση Επίτροπε Γιώχανσον. Εδώ σε αυτή την Επιτροπή αναφέρατε τη σημασία του να εφαρμοστούν όσα ήδη έχουν ε, εγκριθεί και ότι πρέπει να υπάρχει με βέβαια εμπιστοσύνη ώστε να υπάρξει στενή συνεργασία για τις κοινέ απειλέ ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας μεταξύ των οποίων του οργανωμένου εγκλήματος και της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε και αυτό σήμερα. Σε ό,τι αφορά το μέλλον τη εσωτερική λοιπόν ασφάλεια και τη στρατηγική μα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν ήδη έχετε εντοπίσει νέα μέτρα για να δείτε ποιε είναι οι, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του βίαιου οργανωμένου εγκλήματος. Λόγω χάρη πώς θα αντιμετωπίσετε την εμπορία ναρκωτικών, ε, μια από τις βασικότερες πηγές εσόδων για αυτές τις ομάδες. Και ακόμα μια ερώτηση αφορά έναν άλλο τομέα που για μένα είναι σημαντικό, είναι ο τομέα της διακίνηση. Διότι το είπατε και στην εισαγωγή σα. Το άκουσα και νωρίτερα. Ο ε, συντονιστής της καταπολέμησης της διακίνησης ε, θα καταργηθεί ως θέση. Γιατί ξέρουμε ότι η εμπορία έχει αυξηθεί δραματικά. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μέκερ. Δεν τον βλέπω βέβαια στην αίθουσα. Κυρία Γκαρθαουμπουντούα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιώχανσον, στην τελευταία έκθεση του Οκτωβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας μιλούσε για, αναφερόντουσαν στόχοι για εκείνα τα παιδιά που γυρνούν από περιοχές ε, συγκρούσεων ε, στις οποίες λειτουργούσε το ISIS και τα οποία είχαν ε, ριζοσπαστικοποιηθεί και ασκήσει βία. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε τι έχει γίνει, πόσοι από αυτούς τους στόχους έχουν ε, υλοποιηθεί, έχει, έχουν γίνει αυτά τα workshop τα οποία είχαν ανακοινωθεί, έχουν μεταδοθεί σχετικές, τα σχετικά συμπεράσματα στα κράτη-μέλη. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτές τις περιοχές οι άνθρωποι αυτοί έχουν ε, υποστεί μια πλήση εγκεφάλου. Και δεν πρόκειται λοιπόν για τη μετάδοση των, των μηνυμάτων υπέρ της τρομοκρατίας και της βίας μόνο μέσω του ίντερνετ, θα πρέπει να δούμε και τους άλλους διάβλους. Ο κύριος Σεβάιμερ, ε, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, κυρία Επίτροπε. Στη στρατηγική ασφάλειας που ισχύει για ε, το διάστημα 2015 έως 2020 αναφέρεται ο βίαιος εξτρεμισμός. Όταν λοιπόν κύριε Επίτροπε μιλάτε για τους προβληματισμούς γύρω από την ε, τρομοκρατία, πάλι μιλάτε με γενικούς όρους. Μιλάμε για τρομοκρατία, ριζοσπαστικοποίηση, ε, ε, τζιχαντιστές ε, τρομοκράτες, τρομοκράτες ριζοσπαστικοποιημένους ε, στις χώρες τους. Τα τελευταία 8 χρόνια μιλάμε κυρίως για τον Ισλαμικό για, για την Ισλαμική τρομοκρατία και τον Σαλαφισμό. Ρωτώ λοιπόν, είσαστε διατεθειμένοι να φροντίσετε να δοθεί τέλος στις ε, διατυπώσεις αυτές ε, και να ε, έχουμε πιο σωστή διατύπωση, πιο σωστή ορολογία στο θέμα αυτό. Κύριε Πιόρκ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω το εξή. Ε, είπατε, κυρία Επίτροπε, στην εισαγωγή σας ότι υπάρχουν πολλές ε, πτυχές, ε, προσωπική ακαιρεότητα, αξιοπρέπεια, ισότητα απέναντι στον νόμο. Βλέπουμε πολλή βία εις βάρος των γυναικών, ομοφοβία και να γίνεται κανονική πια η βία στον δημόσιο χώρο μεγάλες βάσεις δεδομένων ε, προβλέπεται να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες ε, και να ε, συγχωνευτούν. Εγώ βλέπω να υπάρχει εδώ ένα τεράστιο κενό που ζητώ από εσά να κλείσετε. Θα πρέπει όλα αυτά να βασίζονται στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, στον επόπτη προστασίας δεδομένων και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τι σχέδια έχετε όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, ώστε ε, να μην υφιστάμεθα βία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή προς τις γυναίκες σήμερα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Όπως ξέρετε, ο Η Ισλαμική τρομοκρατία είναι απειλή για, τους, ε, για την εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Καλωσορίζω τι δηλώσει σα και αυτέ τι περασμένε εβδομάδε κυρίω την επικυροποίηση τη εντολή τη Europol. Βρίσκω το θέμα αυτό είναι κέριο και θα πρέπει να ε, ξεχρονίσουμε και την πολιτική μα κατά τη τρομοκρατία. Ωστόσο, ελπίζω ότι αυτέ είναι απλώ οι πρώτε πρωτοβουλίε που θα δούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα βήματα, γιατί θα χρειαστούμε πολύ περισσότερα. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να πείτε δύο λόγια για το αν σκοπεύετε να προβλέψετε νεότερες πρωτοβουλίες για τον εξυγχρονισμό του ορισμού α, ε, του οργανωμένου εγκλήματος, λόγω χάρη, ε, μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχει δηλαδή ένας κοινό και να είμαστε πιο συνεπείς. Επίσης, πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση από τρίτες χώρες των τρομοκρατικών ενεργειών στην Ευρώπη. Αυτό είναι πραγματική απειλή για τη δημοκρατία μας. Και οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα θα ήταν ευπρόσδεκτη. Κυρία Τζόντσεβα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μόλις μας δώσατε. Χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση. Πρέπει να δούμε όμως και τι στατιστικές χρειαζόμαστε και τους απαραίτητους πόρους. Από όσα έχω δει ως τώρα, αμφιβάλλω για το αν η Europol και το Κολέγιο μπορούν να προβλέψουν ε, τις απαραίτητες δράσεις για το πρόγραμμα που θέλετε να προτείνετε. Κυρίως πρέπει να δούμε και την διαφθορά ως ένα τομέα προτεραιότητας παντού ξεπηδάει σε όλα τα θέματα ω ένα ε, σαφή κίνδυνο. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε το θέμα αυτό. Την περασμένη εβδομάδα η Transparency International ήδη σε μια έκθεσή τη αναφέρει ότι η κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη επιδεινώνεται. Και στη δική μου χώρα μεταξύ άλλων, ε, στη Βουλγαρία. Ε, εδώ και κάποια χρόνια οι δυσκολίες που προκαλεί η διαφθορά έχουν υποτιμηθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ λίγα τα ευρωπαϊκά εργαλεία που διευθετούν το χώρο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπονήσει μια σφαιρική στρατηγική κατά της διαφθοράς. Είναι η στιγμή να γίνει μια αλλαγή. Ευχαριστούμε η κυρία Κελέα. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Ήθελα να σχολιάσω την αναφορά σας στην Europol. Τονίσατε την ανάγκη να ενισχυθεί η εντολή τους. Πράγματι, μεγαλύτερη και περισσότερη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών είναι απαραίτητη. Θα ήθελα εδώ να επικαλεστώ ε, ε, την ε, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού FBI με συγκεκριμένους στόχους, ίσως με κάποιες μεταβατικές φάσεις, για να υπάρξει αποτελεσματικότερη αστυνομική συνεργασία και να αντιμετωπίσουμε τις ε, απειλές που διαρκώς μεταβάλλονται και που είναι διασυνοριακές, τα διαπερνούν τα σύνορα. Μιλήσατε για το ψηφιακό τομέα, αλλά οι μορφές εγκληματικών ενεργειών που βλέπουμε, είτε μέσω προσώπων, είτε μέσω επιθέσεων, είτε μέσω δράσεων παρανόμων όπως την ε, διακίνηση ναρκωτικών ξεπερνούν τα σύνορα. Βλέπουμε ε, και οι μαχητές, οι ξένοι μαχητές που επιστρέφουν να είναι μια απειλή και εκείνοι διασχίζουν τα σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν να μας πείτε λίγο περισσότερα για τις πρωτοβουλίες σας στον τομέα αυτό για να γίνουμε δυνατότεροι μαζί με μια ε, δυνατή αστυνομία που θα μπορεί να μας προστατεύσει. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπρέιερ για τους πρασίνους. Ένα λεπτό. Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ θετικά στην πρότασή σας για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία από τρομοκράτες που έχουν ε, μεγαλώσει στην Ευρώπη και την εμπορία των παράνομων πυροβόλων. Ήθελα επίσης να αναφέρω ότι δεν σχολιάσατε την πρόταση για την τήρηση δεδομένων. Και αυτό είναι θετικό. Πολύ καλά κάνατε γιατί είναι φοβερή παρεμβολή στον ιδιωτικό βίο όλων και στο απόρριτο στο οποίο όλοι έχουμε δικαίωμα. Ε, όμως ε, πολλές νέες προτάσεις με ανησυχούν, όπως οι προτάσεις για μέσα παρακολούθησης και εποπτείας. Η Επιτροπή μας πριν από λίγες εβδομάδες ζήτησε να επικεντρωθείτε στην ε, υλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, αντί να περάσετε στην υποβολή νέων προτάσεων. Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές και τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και την κρυπτογράφηση. Τι ακριβώς προτείνετε, δεν το πολύ κατάλαβα. Ε, γιατί η κρυπτογράφηση ε, προστατεύει τους πολίτες από την κλοπή της ταυτότητάς τους, τις τρευλώσεις, την ε, παράνομη παρακολούθησή τους. Μην τα περιγράφετε σαν εργαλεία για τους εγκληματίες μόνο και καλλιεργείτε τον φόβο για να δημιουργήσετε τέτοιες προσδοκίες. Κύριος Μπουσάρα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε για την πρώτη σας παρουσίαση Αναφερθήκατε ήδη από στην πρώτη σας παρουσίαση στο γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό επαναπροωθήσεων και ε, επιστροφών. Συγγνώμη. Ε, θα ήθελα να πείτε τι κάνουμε για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Πώς προχωρούν οι, οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο, με την Αλγερία για συμφωνίες επανεισδοχής. Επίσης, τον Ιούνιο του 2018 είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων η Επιτροπή θα βοηθούσε στη δημιουργία περιφερειακών πλατφορμών. Σκοπεύετε να προωθήσετε αυτό το μοντέλο για πλατφόρμες τις οποίες θα μπορεί κανείς στην τρίτη χώρα να υποβάλει έτοιμα ε, ασύλου έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε με αυτόν τον τρόπο την εμπορία ανθρώπων. Ε, μετά, Brexit και είναι προφανές ότι το Γιβραλτάρ είναι ένα ε, μια περιοχή στην οποία υπάρχει δραστηριοποίηση διεθνών εγκληματικών ομάδων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διακίνηση. Έχει τη διάθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξανανοιξει αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Βαρέρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα γνωρίζετε ότι στη χώρα των Βάσκων προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το γεγονό ότι η ερευνητική διαδικασία έθεσε τέλος στην ε, βία και ότι η... θα ήθελα να επιθυμίσω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2017 για τα συστήματα των φυλακών, όπου μεταξύ άλλων καταδικάζει την πολιτική ε, ορισμένων κρατών μελών για κράτηση απομόνωση και επίσης την πολιτική τους να στέλνουν τους κρατούμενους σε φυλακές μακριά από το χώρο διαμονής της οικογένειάς τους. Πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να βοηθήσουν στην υλοποίηση της πολιτικής της ειρηνευτικής στην περιοχή της χώρας των Βάσκων. Έχει κάνει οτιδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ζητήματα αυτά από, από τότε που πέρασε αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Κέρναρ. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Ήδη έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στη Δανία τις τελευταίες εβδομάδες με διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είπατε ότι θα χρειαστεί νομοθεσία και δομημένος διάλογος με την Επιτροπή μας. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό το σκάνδαλο το πρόσφατο θα αλλάξει την θέση σας και με ποιον τρόπο αξιολογείται τα υφιστάμενα καθεστώτα για την διατήρηση δεδομένων και για το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υλικό. Εγώ πιστεύω ότι τα υφιστάμενα συστήματα είναι επαρκή και δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Και επίσης, σκοπεύεται να επεκτείνεται το σύστημα PNR. Οι Υπουργοί Εσωτερικών προσπαθούν και πιέζουν να επεκταθεί το σύστημα PNR της διατήρηση προσωπικών δεδομένων των επιβατών, εκτός από τα αεροπλάνα και σε άλλες μεθόδους μεταφορέ, όπως για παράδειγμα τα τρένα. Ποια είναι η θέση σα γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι μετά την τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή στο Ιράκ και στη Συρία, παρόλο που φαίνεται να έχει νικηθεί σε ορισμένε περιοχές το ε, ε, το ISIS συνεχίζουν συνεχίζουμε να ανησυχούμε για το γεγονό ότι έχουν παραμείνει κάποιοι μαχητέ, οι οποίοι βρίσκονται σε Συριακέ και, και Ιρακινές φυλακέ. Το ζήτημα λοιπόν της, ε, του επαναπατρισμού ε, ορισμένων παιδιών που ίσω ε, έχουν ρίζος παστικοποιηθεί είναι, είναι ουσιαστική σημασία. Πώ θα φροντίσουμε για την ασφάλεια των πολιτών μα, εάν επαναπατριστούν τέτοια άτομα με πιθανώς ένα επικίνδυνο προφίλ και πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε εκ των προτέρων να γίνεται μια ταυτοποίηση του προφίλ ενός προσώπου που μπορεί να, θέτει, να, να, να αντιπροσωπεύει κίνδυνο. Για η κυρία Μπρίκμο, για ανθρωπιστικού χαρακτηρα ζητήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με την επαναπρόθεση, τον επαναπατρισμό των παιδιών τζιχαντιστών. Τι θα κάνετε για τη συνεργασία των κατώμελων σε αυτό το τομέα και ακούσαμε από τις διωτικές αρχές, από τις διαδικαστικές αρχές, τι αρμοδιότητες πρέπει να αναλάβουν στην επαναπρόθεση, ώστε να βεβαιωθούν ότι οι ξένοι μαχητές, οι ε, τζιχαντιστές, δικάζονται στις δικές μας τις χώρες για να μπορούμε να ελέγξουμε λίγο τα πράγματα και να είμαστε βέβαιοι ότι οι ποινές τους θα είναι πραγματικές ότι δεν θα επανέλθουν σε αυτό που έκαναν πριν. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κυρία Επίτροπε, και για τη μεταναστευτική πολιτική. Δεν πιστεύετε ότι μια μεταναστευτική πολιτική που αναφασίζεται στα ρουπνά δικαιώματα, την υποδοχή, την αλληλεγγύη και τι νόμιμε οδού που επιτρέπουν να έρθει ο κόσμο στην επικρατεία μα θα επέτρεπε να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων και θα διασφάλιζε δικαιώματα στον κόσμο, ιδίω του μετανάστε που σήμερα είναι πραγματικά θύματα τη εμπορία αλλά και τη επισφαλού θέση στην οποία βρίσκονται, να προσπαθούν να διασχίσουν ολόκληρε υπήρου αλλά και τα σύνορα Ευχαριστούμε. Κέμπε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, έχω μια ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψης. Γνωρίζουμε ότι αυτό ήταν ένα αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, ωστόσο ε, τώρα πια δεν ε, εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες για πολιτικούς λόγους μη κατανοητού για εμάς. Αυτό ισχύει στην περίπτωση υπόπτου που δεν εστάλει στην Πολωνία. Σκοπεύεται να ενισχύσετε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη ώστε πάντα να ε, εφαρμόζεται. Και επίσης ε, πώς βλέπετε εσείς ε, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2015 για την μετανάστευση για το διάστημα 2015-2020. Η στρατηγική αυτή έχει παίξει το ρόλο της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εκπονήσει νέο σχέδιο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την επιστροφή ε, πολεμιστών ε, Ισλαμιστών. Ε, τι μέτρα σκοπεύετε να υιοθετήσετε για να εμποδίσετε την επιστροφή τέτοιων προσώπων και των οικογενειών τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό μόνο, κυρία Κινίτση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο για την ε, διαθεσιμότητά της να, περάσουμε σε διάλογο. Για το οργανωμένο έγκλημα που όλο ένα πλώνει τις ρίζες της στην επικράτειά μας και παρεμβαίνει στο χρηματοπιστωτικό μας ε, σύστημα και τα οικονομικά των χωρών μας με τη διαφθορά, την... Ε, το ξέπλυμα και τις απάτες. Πρέπει για να αντιμετωπίσουμε δραστικά το οργανωμένο έγκλημα να έχουμε καλύτερη αναχέτηση με καλή ανταλλαγή πληροφοριών και την τήρηση δεδομένων που να είναι αποτελεσματική. Σα ρωτώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά τι έρευνε για την καταπολέμηση του ξε... κυρίω κατά του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Ε, κυρία Επίτροπε, λέτε ότι θα πρέπει να εντοπίζονται ύποπτε συναλλαγέ και να υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων μέχρι των αρμόδιων αρχών. Θεωρείτε όμω ότι για την ώρα είναι αρκετά όσα γίνονται, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να υπάρχει ταχύτερη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων για τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές των κρατών μελών ακόμη και με την έγκριση και την υποστήριξη της Europol. Και επίσης φρονείται ότι μπορεί να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο των αρχών κατά της διαφθοράς για να ε, μπορέσουμε να καλύψουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν στη συλλογή δεδομένων στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα, κυρία Επίτροπε Ιωάννησον. Αντιλαμβάνομαι ότι το να προσπαθήσετε να απαντήσετε και να συνοψίσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι δεν θα είναι εύκολο. Βέβαια έχετε και τις δύο βοηθούς σας που σας επικουρούν και εκ των προτέρων θα πω ότι θα εκτιμήσω την προσπάθεια που θα κάνετε γιατί είναι πολλές αυτές οι ερωτήσεις αλλά έτσι είναι αυτή η δουλειά. Τα θέματα της αρμοδιότητας σας ενδιαφέρουν προφανώς πολύ τους συναδέλφους. Και θα σας δώσω λοιπόν το λόγο για να ακούσουμε τις απαντήσεις σας σε όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύ καλή προσπάθεια που πιστεύω ότι θα κάνετε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις και για πολλές από αυτές τις ιδέες που υποβάλλατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν κάτι μου διαφύγει, ευχαριστώ να επανέλθω, γιατί ορισμένα από αυτά μάλιστα είναι θέματα που καλύτερα να τα συζητούμε διαρκώς. Πρώτα απ' όλα, Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, κυρία Μέτσολα. Αυτό είναι μέρος της νέας συμφωνίας για το άσυλο και τη μετανάστευση που θα προτείνουμε. Ένα σημαντικό στοιχείο. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο χώρος έγκαι δεν προστατεύεται όπως θα έπρεπε. Γνωρίζουμε ότι θα έπρεπε να υφίστανται συστηματικοί έλεγχοι και αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από μελέτες, που δείχνουν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να ξεφύγουν και να περάσουν από τους συνοριακούς ελέγχους χωρίς να ελεγχθούν. Ε, ένα ποσοστό της τάξης του 22% αναφέρεται. Επομένως, τίθεται ένα θέμα εφαρμογής της νομοθεσίας και πώς κανείς ακολουθεί τους κανόνες που έχουμε ήδη θεσπίσει για να ε, ε, ενισχύσει την έλεγχο των εξωτερικών συγχωνόρων, που το θεωρώ κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών. Όπως είπατε, η διαλειτουργικότητα εδώ έχει κρίσιμο χαρακτήρα. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ροή, σωστή ροή δεδομένων από και προ κάθε κράτο μέλο. και επίση και εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και με τι υπηρεσίε τη Επιτροπής. Κυρία Σίπελ και κυρία Ίντφελτ τονίσατε τη σημασία της εφαρμογής. Και σε αυτό συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Θα επιδιώξουμε 100% να εφαρμόζονται οι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό. Όμως δεν βλέπω να είναι αντικρουόμενο το να επιδιώξουμε ταυτόχρονα να έχουμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ή επικυροποίηση παλαιάς νομοθεσίας. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί στενή ε, συνεργασία και η ιδέα σας για να φτιαχτεί ένα scoreboard, ένα βαθμονόμιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ε, δικαιοσύνης θα είναι μια καλή ιδέα. Θα την εξετάσω. Επίσης θα ήθελα να καλύψει το πρόγραμμα Εράσμους και τις αστυνομικές αρχές ή γενικότερα τις διεκτικές αρχές. Αυτό ίσως είναι κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε προγράμματα τα οποία ήδη υφίστανται και για τους αξιωματικούς των διοκτικών αρχών για να εκπαιδεύει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι επίσης κάτι που εξετάζω. Για το ζήτημα τώρα της βίας κατά των γυναικών που το ανέφερε η κυρία Ιντφελτ και η κυρία Γιώργεν και άλλοι, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Οι γυναίκες και τα παιδιά δεν είναι ασφαλείς στα, στις οικίες τους, στην οικογένειά τους. Και εκεί είναι το πρόβλημα και ε, επ' αυτού θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Βεβαίω αυτό είναι κυρίω ζήτημα των εθνικών αρχών, αστυνομικών και δικαστικών. Αλλά οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να τι βοηθήσουμε, θα το πράξουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση με τη συνάδελφο Ελένα Ντάλη, η οποία είναι υπεύθυνη ω επίτροπο για τα ζητήματα ισότητα. Γιατί ε, σκεφτήκαμε ίσω κάποια πράγματα να μπορέσουμε να τα αναλάβουμε ω πρωτοβουλίε από κοινού. Στη Europol, για τη Europol, πιστεύω ότι χρειάζεται να επικυρωποιήσουμε την εντολή τη, με βάση επίσης την εντολή που τη δίνεται με την απόφαση πριν, είναι σημαντικό όλες αυτές οι εντολές αυτών των υπηρεσιών να μην γίνονται παροχημένες. Αλλά έχετε δίκιο ότι και το ζήτημα του προπολογισμού είναι σημαντικό. Το αναφέρατε πολλοί από εσά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την Europol, γιατί τις έχουν αποδοθεί περισσότερα καθήκοντα και έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εδώ. Γιατί η κυρία Στίκ Πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύονται αυτά. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ισότιμοι κανόνες οι ε, ισότιμοι κανόνε είναι προαπαιτούμενο για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Ότι, ε, να μπορούμε δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι έχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το επιδιώξουμε. Για το νέο θεματολόγιο για τα ναρκωτικά. Δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε στα θέματα στα οποία τα κράτη-μέλη είναι διχασμένα είναι καλύτερα να εστιάσουμε σε εκείνα από τα θέματα στα οποία διαπιστώνουμε ότι θα υπέρξουν ωφέλη από τη συνεργασία. Για τη διασυνοριακό έγκλημα. Βεβαίως χρειάζεται καλύτερη συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται καλή προστασία προσωπικών δεδομένων, συστήματα τα οποία να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους διαλειτουργικά και να επιτρέψουν στις διαφορετικές αρχές να συνεργάζονται. Για το ζήτημα της έρευνας. Και αυτό είναι σημαντικό. Σκέφτεται η Europol να ξεκινήσει να ανοίξει ένα εργαστήριο καινοτομία για να μελετάει αυτό πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε νέες μορφές απειλών και πώς μπορούν οι διακτικές αρχές να τις αντιμετωπίζουν αυτές τις νέες απειλές. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ιδέα που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Για τη νέα εντολή της Frontex η οποία, θα, η οποία ε, ετέθησε ισχύ το Δεκέμβριο του 2019. Υπό αυτή την εντολή, όπως έλεγα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ε, αυξηθούν οι επιστροφέ εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί το ποσοστό των επιστροφών. Αυτό θα είναι επίση στοιχείο τη νέα ε, Συμφωνία για το άσυλο και τη μετανάστευση. Αλλά ε, πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι μόνο αρμοδιότητα τη Frontex. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και καλύτερε συμφωνίε με τι τρίτε χώρε, έτσι ώστε και εμεί να τι βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τους διακινητές αλλά και να δέχονται να ε, γυρίσουν σε αυτές οι πολίτες τους όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τους αρνείται την παραμονή. Επίσης είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει μια αρνητική, μια απόρριψη του αιτήματο ασύλου να προχωράει γρήγορα η διαδικασία και επίσης χρειάζεται και η Frontex να βελτιωθεί στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει στην πράξη τις απελάσεις για το σύστημα Schengen, συγγνώμη, για το πληροφοριακό σύστημα Schengen, το ΣΥΣ, το οποίο α, έτυχε κατάχρησης, είναι σκάνδαλο, είναι απαράδεικτο, είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν, ελπίζω, θα υπάρξουν μάλλον, ελπίζω, συστάσεις του Συμβουλίου σχετικές και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το λάβουμε υπόψη μας και στην νέα διαπραγμάτευση με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία γνωρίζει ότι θα είναι με ένα πάρα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα για να δούμε ποιε θα είναι οι σχέσει μα με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά Brexit και το ζήτημα της ασφάλειας, ε, μια διαπραγμάτευση που μπορεί να συνεχιστεί και μετά το Δεκέμβριο, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα το παρακολουθήσω στενά. βεβαίω, ο Μισελ Μπαγνιέ είναι αρμόδιος για το σύνολο της διαπραγμάτευσης, αλλά ως αρμόδια για τα ζητήματα της ιστορικής ασφάλειας, Βεβαίω θα συμπροεδρεύω και θα προσέχω και θα παρακολουθήσω στενά αυτό το σκέλος της διαπραγμάτευσης. για το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η κυρία Βασιλιάδου, η τρέχουσα συντονίστρια πολέμηση του τράφικινγκ, ήταν εξαιρετική και ελπίζουμε να ε, συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά από ό,τι έμαθα δεν επιτρέπεται εξαιτία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας να παραταθεί η θητεία της περισσότερο. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία επιλογή ε, ενό άλλου ατόμου. Το λυπάμαι γιατί είναι εξαιρετική και έκανε πολύ καλή δουλειά. Ελπίζω να βρω, θα προσπαθήσω να βρω μια λύση, αλλά δεδομένη τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και των κανόνων χρειάζεται να ξεκινήσει μια εξωτερική διαδικασία επιλογή. Για να συνεχιστεί αυτό. Ναι. Ναι, απάντησε η Επίτροπη σε σχόλιο εκτό μικροφώνου, θα μπορούσε να είναι η ίδια. Πρόεδρος ήθελα να το επισημάνω κι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε, ήταν στη, ε, στη θέση αυτή στην προηγούμενη εντολή να είναι υποψήφιο για την επόμενη εντολή. Απάντηση τη Επιτρόπου. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Η θέση θα υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία στην οποία η, ίδια θα μπορούσε να υποβάλει υποψηφιότητα. Αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα επιλεγεί. Αυτό που σας λέω είναι ότι δεν μπορούμε αυτομάτως να παρατείνουμε τη θητεία της, γιατί έχει ήδη συμβεί αυτό, έχει φτάσει σε ένα σύνολο 9, 9 θητείας. Ε, με βάση την νομοθεσία πρέπει να ανοίξει πάλι θέση. Τώρα, για τους ξένους μαχητές... Ε, Θα επανέλθω γιατί πολύ θέσατε το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτό είναι μια εθνική απόφαση. Είναι, στην, είναι κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέξουν εάν θα δεχτούν αυτά τα πρόσωπα, εάν θα ε, ακολουθήσουν κάποια ε, διαδικασία έρευνας και ποια, τι θα κάνουν. Από την πλευρά μας, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για παράδειγμα, θα μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε για να συλλέξουν αποδεικτικό υλικό εάν επιθυμούν να πάνε σε δίκη. Ή μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ τους. Θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε ε, ε, τις, τις, τις δραστηριότητές τους, αλλά είναι εθνική αρμοδιότητα να αποφασίσουν τι θα πράξουν με τα πρόσωπα αυτά. για αυτόν τον εξτρεμισμό που οδηγεί σε πράξεις βίας. Είναι κατά την άποψή μου απαραίτητο να συμπεριλαμβάνουμε όλες τις μορφές του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας που απειλούν τους πολίτες μας. Όπως είπα, η τζιχαντιστική τρομοκρατία παραμένει μια απειλή, αλλά και η ακροδεξιά τρομοκρατία και βία έχει αρχίσει να αυξάνεται και παραμένει μια απελή. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να τα θεωρούμε αυτά τα δύο ως δύο άκρα και να τα αντιπαραθέτουμε, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και τα δύο. Με ρωτήσατε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για τα δικαιώματα των γυναικών. Το, αναφέρατε ήδη και εσείς. Το θέμα δεν είναι να αντιμετωπίζει μόνο τα εγκλήματα κανείς στο ίντερνετ, online, αλλά το θέμα είναι για να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γνωρίζετε ότι η αρμοδιότητα τη ανάληψη μια δράση ή τη δίωξη είναι εθνική αρμοδιότητα. Το θέμα είναι να δούμε πώ μπορεί να βοηθήσει αυτέ τι αρχέ τι διοκτικέ η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχε τη ιδιοκτικε η ευρωπαικη ενωση η να, ε, ε, να, να, να συνεισφέρει περισσότερο όταν υπάρχει διασυνοριακό έγκλημα, γιατί εκεί πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω. Κύριο Σταμπέο, νομίζω ανέφερε την χρηματοδότηση από τρίτε χώρες του, ε, της εξτρεμιστικής ε, βίας και τρομοκρατίας. Είναι σωστή η παρατήρησή σας και θα την εξετάσω περισσότερο. Ε, τώρα για το ζήτημα του αν χρειαζόμαστε εναρμονισμένους ορισμούς, εδώ πιστεύω πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όταν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε την ομοθεσία μας. Αλλά είναι να προσέξουμε να μην σπαταλάμε την ενέργειά μας σε κάτι στο οποίο δεν είναι πραγματικά απαραίτητο, εάν πραγματικά δηλαδή δεν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Η διαφθορά είναι ένα πρόβλημα ε, υφιστάμενο, γνωστό, και έχει πλέον θεωρηθεί ένα πολύ μεγάλο σημαντικό στοιχείο της, του κράτους δικαίου που έχει γίνει πια σημαντική ε, προτεραιότητα που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, το εάν θα ξεκινήσουν διαδικασίες ε, επί δεν μπορώ να το αποκλείσω εάν χρειαστεί. Για τι επιστροφέ, εντάξει νομίζω ήδη απάντησα ότι, ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε πολλού τομεί Για τη διατήρηση δεδομένων. Όπως γνωρίζετε, η οδηγία για την διατήρηση προσωπικών δεδομένων ακυρώθηκε. Επομένως, αυτό θα πρέπει να ευληφθεί υπόψη και θα πρέπει να σκεφτούμε αν χρειαστεί να προτείνουμε μια νέα οδηγία. Εκκρεμούν υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει υποβάλει προτάσεις για τις ε, ε, υποθέσεις αυτές Επομένως, περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Και ανάλογα με τις αποφάσεις του δικαστηρίου θα εξετάσουμε κατά πόσο χρειάζεται νέα νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή ή όχι. Για το PNR κάνουμε αυτή τη στιγμή μια αξιολόγηση. Θα παρουσιάσουμε δηλαδή μια αξιολόγηση της τρέχουσας νομοθεσίας, θα την παρουσιάσουμε το Μάιο και επί τη βάση αυτή θα σκεφτούμε αν χρειάζεται να φέρουμε νέε προτάσει ή όχι. για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο και την καταπολέμησή του. Ε, είναι επίση σημαντικό και είναι ένα από του λόγου για τον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η έντολη τη Europol για να μπορεί να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών για τα θέματα αυτά. Αλλά εδώ υπάρχει και συντρέχουσα αρμοδιότητα του Επιτρόπου Ρέιντερ. Επομένω, ε, η όποια πρόταση μάλλον από κοινού θα έρθει. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε Ιωάννσον. Ευχαριστούμε τους διερμηνείς, διότι τους ζητήσαμε λίγο χρόνο παραπάνω και το πρωί και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ, λοιπόν. Ε, δεν είχαμε χρόνο να καλύψουμε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Νομίζω όμως ότι αρκεί για τώρα αυτό, αυτή η ανταλλαγή απόψεων και ο διάλογος που είχαμε με εσάς, κυρία Επίτροπε, ε, δώσαμε την ε, δυνατότητα στους ε, βουλευτές να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ακόμη και αν είναι θέματα ε, που ε, ανήκουν σε αρμοδιότητες αλληλού. Πάντως σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα αυτή ε, και Προσβλέπουμε στη συνέχιση του στρατηγικού αυτού διαλόγου με την Επίτροπο πάνω σε θέματα εσωτερικών και ασφάλειας. Σας ευχαριστώ και πάλι.